να ζητήσει έκδοση του δημοσιογράφου αυτού ή η τουρκια ή να τον συλλάβει ή να τον απάγει. Ε, τι θα πείτε τότε. Επειδή λέει παραβίασε ε, τα, τα μυστικά του Ιράν, της Τουρκίας ή οτιδήποτε. Μην παίζετε τον Ποντιοπιλάτο λοιπόν εδώ πέρα όταν κινδυνεύει η ελεύθερη πληροφόρηση και σταυρώνονται οι ε, καταγγέλλοντες. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από την Άννα Γκόμες. Την δέχεστε, ναι. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκόμες. Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Είμαστε πολιτικό σώμα και μπορούμε να εκφέρουμε πολιτική κρίση. Και αυτό κάνουμε. Λέμε δεν πρέπει να εκδοθεί στη ΣΥΠΑ από την άλλη αναμένουμε τα δικαστήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο που ευτυχώς ε, θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, δεσμεύονται από την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις ε, συνθήκες και άρα υπάρχει κάποια νομική και όχι πολιτική βάση για να μην υπάρξει έκδοση σε μια χώρα που έχει ακόμα θανατική ποινή. Συμφωνείτε κύριε Κουλούγλου. Make... Συμφωνώ πλήρω. Πρέπει να κάνουμε μια δήλωση. Έχουμε κάνει δηλώσει επιδηλώσεων για τη Βενεζουέλα, την Τουρκία, ε, ε, για τα πάντα. Και ο συναδελφός μου εκεί πέρα μιλάει για νομική διαδικασία. Έγινε σεβαστή η νομική διαδικασία στην περίπτωση άλλων χωρών. Κάνουμε παρεμβάσεις δηλώσεις. Γιατί όχι τώρα. Επειδή είναι σε αυτό το χάλι η Βρετανική κυβέρνηση λόγω Brexit και προσπαθεί να ξεμπλέξει με τον αντιπεριστασμό του Ασάζ. Δεν είναι σωστό αυτό. Όχι. Είστε πολιτικός, πρέπει να λάβετε μια θέση. Είστε υπέρ ή κατά της έκδοσης. Σας ευχαριστώ ε, βεβαίως ε, ερωτηθήκατε, έχετε δικαίωμα να απαντήσετε. Κυρία Πρόεδρε, ε, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω. Είναι νομικό ζήτημα. Αυτό είναι. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, τώρα, εάν είστε υπέρ του οι πολιτικοί να παρεμβαίνουν στις δικαστικές διαδικασίες, είναι κάτι το κατανοητό και θεμητό. Αλλά εγώ ε, δεν συμφωνώ. Αλλά είναι δικαίωμά σα. να το υποστηρίζετε αυτό. Αλλά είναι τελείως αντίθετο με τον τρόπο που ε, λειτουργούν οι δυτικές δημοκρατίες. Η διάκριση της εκτελεστικής από τη δικαστική εξουσία είναι θεμελιώδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα Μιράντα για ένα λεπτό, εκ μέρους των Πρασίνων. Ένα λεπτό σας δίνω το λόγο. Θα σας ρωτήσω το εξής, συνάδελφε. Τι γίνεται με τις δίκες στην Τουρκία. Η Τουρκία σωστά λέει ότι αυτό είναι νομικό ζήτημα, νομική, νόμιμη δράση και ότι πρέπει να σεβαστούμε τη, νόμιμη, τη νομική διαδικασία στην Τουρκία και να μην παρέμβουμε τότε γιατί εμείς κάναμε τόσες δηλώσεις κατά δικών στην Τουρκία. Γιατί. I keep this as a Ρητορικό το θεωρώ το ερώτημα. Επιθυμείτε να απαντήσετε. Όχι, ναι. Να απαντήσω σε μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό που προτείνει, διατείνεται ο συνάδελφος, είναι ότι η Βρετανική κυβέρνηση θα έπρεπε να παρέμβει σε μια δικαστική διαδικασία στην Αγγλία. Αυτό που λέτε για την Τουρκία είναι να παρέμβετε ή να επιδιώξουμε να παρέμβουμε στην Τουρκία. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ με τις επικρίσεις κατά της Τουρκίας. Και μακάρι η κυβέρνησή μου και άλλες κυβερνήσεις να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία ποτέ δεν θα γίνει μέλος, τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μέλος ή όχι. Ευχαριστώ συνάδελφοι και οι δύο πλευρές ακούστηκαν. Θα μπορούσατε να πιάσετε μεγάλη κουβέντα. Ας δώσουμε το λόγο στην επόμενη συνάδελφα Άννα Μιράντα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Την ε, Δευτέρα είχα ραντεβού με τον ε, Ζουλένα Σάνς ε, στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο. Δεν πήγα γιατί στο μεταξύ συνελήφθη. Παραβιάστηκε το δικαίωμά του σε άσυλο και φυλακίστηκε. Ε, το δικαίωμα του ασύλου σημαίνει προστασία από την θανατική ποινή και απόλυτη προστασία δικαιωμάτων. Το άσυλο που ζήτησε ο Ασάζ είναι για να προστατευτεί από την ε, ηλεκτρική καρέκλα και να προστατευτεί το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας σε μια χώρα που δεν θα είχε δικαίωμα σε δική δίκη. Ε, Παρ' όλα αυτά παραβιάστηκε το δικαίωμα ασύλου του Ζουλιάν Ασάνζ και παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του. Έγιναν δεκτές ε, ε, δεκάδες δίκη ε, καταδίκη ε, στις αμερικανικές φυλακές. Η Βρετανική κυβέρνηση δεν απαιτεί εγγύηση από τις ΗΠΑ για να μην εφαρμογεί της θανατικής ποινής γιατί στις επιστολές που βρέθηκαν στο, στο στην, ε, στην Υπουργή Δικαιοσύνη του Ισημερινού διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν αναλυθεί ούτε εγγυήσει ούτε υποσχέσει να μην εκδοθεί ο Ζουλένα Σαν στι Ηνωμένε Πολιτείε. Το Ηνωμένο Βασίλειο ουδέποτε δεν έδωσε εγγύηση για μη έκδοση. Και θεωρούμε ότι ο σημερινός με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο συντονίστηκαν για να συλλάβουν τον Ασάνζ. Δεν θα πρέπει να εκδοθεί ε, ο Ασάνζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γίνει κάτι τέτοιο οποιοδήποτε δημοσιογράφος που ε, καταγγέλει διαφθορά ή κατάχρηση εξουσίας θα μπορεί να έχει την ίδια μοίρα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Κονέτσνα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα ψηφίσαμε μία οδηγία όπου προβλέπεται η προστασία εκείνων που καταγγέλουν ε, διάφορα γεγονότα και να τους προστατεύουμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε αυτό. Αυτό ψηφίσαμε σήμερα. Σε αυτή την έκθεση και σχετικά με αυτό θα ήθελα να πω ότι όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν ε, τελευταία όπως τα LuxLeaks ή τα Panama Papers Όλα αυτά αποκαλύφθηκαν χάρη σε καταγγέλλοντε. Ήταν προς το δημόσιο συμφέρον. Έτσι δεν είναι. Δεν με νοιάζει πραγματικά. Δεν με νοιάζει αν η Ασάσα Τζούλια Ασάνς είναι προδότης ή είναι ήρωας. Ε, τον θεωρώ σε αυτή τη φάση αυτό το γεγονός δευτερεύουσης σημασίας. Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι ότι αν θέλουμε να προστατεύουμε τους καταγγέλλοντες πρέπει να προστατεύσουμε τον Ασάνς. Θα πρέπει να εκδοθεί προς μια χώρα στην οποία ο πρόεδρος θεωρεί το δημοσιογράφο σαν έναν εχθρό του λαού. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μια τέτοια δικαιοδοσία θα είναι δίκαιη σε μια τέτοια χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο έχει η Επίτροπος η κυρία Γιούροβα. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως. Εμείς ε, ε, υπολογίζουμε πλήρως στην ανεξαρτησία και τον επαγγελματισμό των Βρετανικών δικαστηρίων. Και πιστεύω ακράδαντα ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαίωμα για δίκαιη δύση θα γίνουν πλήρως σεβαστά στις αποφάσεις των Βρετανικών δικαστηρίων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει εκπρόσωπος Ρουμανική Προεδρία, η Υπουργό Τσιότ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, κυρίες και κύριοι, για να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ε, ευκαιρία που μου δώσετε να συζητήσουμε αυτό το επίκαιρο ζήτημα και θα να σας ευχαριστήσω που συζητήσατε αυτό το θέμα της υπόθεσης Ζουλιανασάς και ευχαριστώ για την προσοχή. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, τελείωσε και η ημερήσια διάταξή μας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας αύριο στις 8.30 αύριο το πρωί. Έχει δημοσιοποιηθεί η ατζέντα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ημερήσια διάταξη. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε. Γεια σας.